οι βασικές αρχές που ισχύουν για τον κόσμο ισχύουν και στον τομέα του διαδικτύου ισχύουν μάλλον για τους παρόχους υπηρεσιών. Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο το διαδίκτυο, το κατασκευάσαμε, το εφήβραμε, το ε, εκμεταλλευόμαστε, το χρησιμοποιούμε, αντλούν δηλαδή ωφέλη από αυτό πραγματικοί άνθρωποι. Ε, υπάρχουν απτοί δεσμοί με τον πραγματικό κόσμο. Και σε όλες τις δραστηριότητες όλων των φορέων ε, θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις ίδιες αξίες όπως αυτές που εφαρμόζουμε και στον πραγματικό κόσμο. Πρώτον, ε, τώρα τα θεμελιώδη δικαιώματα που προασπίζουν ε, που προασπίζουμε για, για τους πολίτες πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως και για, στο διαδίκτυο γιατί είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής. Στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωματών δεν έχουμε καμιά υποσημείωση που να λέει εφαρμόζεται αυτό και στο διαδίκτυο ή δεν εφαρμόζεται στο διαδίκτυο. Ε, οι κυβερνήσεις όταν καλούνται να δράσουν για να αντιμετωπίσουν κάποιους από τους κινδύνους στο διαδικτύο, όπως κάνουν και στην ε, καθημερινή ζωή, το θέμα είναι να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Όταν παραβιάζονται δηλαδή τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ιδιωτική ζωή, η ελευθερία της έκφρασης, ε, των σκεφτικών ε, πεπιθήσεων, του συνέρχεστε, Χρειαζόμαστε κριτήρια όπως ε, θεμητή νομική βάση, αναγκαιότητα, αναλογικότητα, ανάγκη περαιτέρω δικλείδων ασφαλείας, Όπως ακούσαμε ήδη, ε, συχνά παραγνωρίζεται αυτό. Θεωρείται δηλαδή ότι το διαδίκτυο σχετίζεται μόνο με ε, νέο τρόπο άσκησης των δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων. Μια νέα ε, παιδική χαρά αν θέλετε. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι Ταυτόχρονα υπάρχουν και νέα χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο και ακριβώς αυτά τα νέα χαρακτηριστικά αποτελούν πρόκληση ε, για την, ε, σε σχέση με την εφαρμογή των παραδοσιακών αξιών του κόσμου στον οποίο ζούμε και το βλέπουμε αυτό μέσα στην έκθεση. Αυτό ο χάρτης δικαιωματών, το Bill of Rights, χρειάζεται ούτω ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναγνωρίσουν την σημασία, να ακολουθούμε τις παραδοσιακέ προσεγγίσεις και στο δικό του τον τομέα ξαναλέω, ε, ας μην ε, το παρουσιάσουμε ως ένα Far West, την Άγρια Δύση, ένα ε, έδαφος που πρέπει να κατακτήσουμε, τέρα incognita. Όχι, απλά υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο το οποίο καλούμαστε να εφαρμόσουμε και στον τομέα του διαδικτύου. Ε, τώρα θα ήθελα... Να σας μιλήσω περισσότερο για το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασία των ατομικών δεδομένων όπως ισχύει μέχρι τώρα. κυρίως στα πλαίσια της οδηγίας 9546. Ε, για την εφαρμοσιμότητα αυτής της οδηγίας ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στον τομέα του διαδικτύου δηλαδή και για όσους δραστηριοποιούνται στο διαδικτύο. Έχουμε και την απόφαση του 10 σε σχέση με την ερμηνεία αυτής της οδηγίας. Υπήρχε μια υπόθεση μιας Σουηδέζας που έκανε θελοντική εργασία στην εκκλησία της και στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας είχε και έναν ιστότοπο με βασικές, πολύ βασικές πληροφορίες. Είναι πολύ παράδοξη αυτή η υπόθεση, αξιοπερίεργη, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση απεφάνθη ως εξής το ΔΕΚ, σαφώς. Ε, η οδηγία είναι εφαρμοστέα και στο διαδίκτυο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το θέμα. Ε, αναφέρονται και κάποια νέα χαρακτηριστικά του διαδικτύου και αναφέρθηκαν κάποιες διατάξεις σε σχέση με την ε, διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών στα πλαίσια του ε, διαδικτύου. Ε, και οι βασικές αρχές οδηγίες είναι εφαρμοστές. Τώρα, ως προς τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχουν τρεις βασικές έννοιες οδηγίες που σχετίζονται με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, ε, το βασικό κομμάτι κατεξοχήν είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, είναι λύει αναφιλεγόμενο το ζήτημα του ορισμού των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Μα αν θεωρήσουμε ότι το διαδίκτυο είναι όπως και ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ε, δεν αλλάζει η αντίληψη περί επεξεργασίας ατομικών δεδομένων. Αλλά η οικονομική, τι γίνεται με την οικονομική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, το business model, ε, το επιχειρηματικό το μοντέλο ε, του διαδικτύου βασίζεται στην αντίληψη ότι είναι ε, πιο ε, στενή η ερμηνεία της έννοιας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και γίνεται μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους ε, κανόνες για την επιγραμμική διαφήμιση παραδείγματο χάνει, online advertising και έχουν τοποθετηθεί και ε, η και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου δημοσίευσε σχάτως μια έκθεση που υποστηρίζει και την ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα ότι όταν μια εταιρεία ε, που δραστηριοποιείται στο ίντερνετ, ε, ένας πάροχος υπηρεσιών, ε, εστιάζει στα ατομικά δεδομένα κάποιου πέραν του ονόματό του, ονοματός του, τόσο περισσότερο μπαίνουμε στο πεδίο των ατομικών δεδομένων. Ξέρετε, ε, δεν μιλάμε για το όνομα και τη διεύθυνση και το τηλέφωνο κάποιου. Μιλάμε για τις διακρίσεις και την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων βάσει κάποιων χαρακτηριστικών τους. Ε, και εγώ το δέχομαι αυτό ότι οι διάφορες δραστηριότητες στο διαδίκτυο βασίζονται στο profiling, ε, δηλαδή στην επιλογή κάποιων και την κατηγοριοποίησή τους μιας την επιλογή μιας ομάδας ανθρώπων. Τώρα δεύτερο θέμα. Ε, στον, ε, στον παραδοσιακό κόσμο έλεγχος της ευθύνη ε, ήταν απλό πράγμα, υπήρχαν δημόσιοι φορείς και από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις. Στο διαδίκτυο υπάρχουν όμως διάφορα στρώματα ευθύνη. Το θέμα της απόδοση ευθυνών ε, είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και όσο πιο περίπλοκο είναι, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνο να εκλείψει η ευθύνη. Ε, και το να αποδίδονται οι ευθύνες ε, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα ε, και γι' αυτό δεν πρέπει να είναι ομιχλώδες το τοπίο στο διαδίκτυο. Δηλαδή, οπωσδήποτε σε αυτές τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα σε όλους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να διευκρινίσουμε ποιος καλείται να υπομειστεί την ευθύνη γιατί. και έχουμε το άρθρο 29, την ομάδα του άρθρου 29 του Ευρωπαϊκού Νομοθέτη να δούμε ακριβώς αυτό το περίπτωμα περίπλοκο περιβάλλον, πώς μπορούμε να εννοήσουμε την, ε, τον έλεγχο και την απόδοση ευθυνών. Τρίτον, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Πρέπει να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Η οδηγία εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και το, ε, μέσα στην οδηγία δίνεται η εξή απάντηση για το εφαρμοστέο δίκαιο, ότι είναι εφαρμοστέα η κείμενη νομοθεσία, εθνική νομοθεσία ε, βάσει της ελεγκτικής αρχής, ε, δηλαδή Εάν κάποιο έχει την έδρα του στη Γαλλία, ένα πάροχο έχει την έδρα στη Γαλλία, τότε είναι εφαρμοστείο το γαλλικό δίκαιο για την επεξεργασία των ατομικών δεδομένων για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και υπάρχει και δεύτερο κανόνα ότι ε, εφαρμόζεται η οικία νομοθεσία όταν χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία μέσα που βρίσκονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους. Ε, πέρα από την περιπλοκότητα του ελέγχου τίθεται και το ζήτημα της έδρας, της εγκατάστασης της εταιρεία. Αλλά αυτό είναι διωγγούμενο πρόβλημα διότι είναι πολύ καλό αυτό από πλευράς απλούστευσης των κανόνων ε, της έννοιας αγοράς, ε, της εσωτερικής αγοράς αλλά θέτει ζήτημα απόδοσης ευθυνών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ε, οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα του εφαρμοστείου δικαίου. Δηλαδή πρώτον να τονίσουμε ποιες είναι οι ε, ισχύουσες αρχές και ενδεχομένως να, ε, να χρειαστεί να μετεξελιχθούν, να διευκρινιστούν, να τις διασαφηνίσουμε. Τώρα, ως προς την ουσία υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Το ένα το συζητήσαμε ήδη, το θέμα της συγκατάθεσης, consent. Μην ξεχνάτε όμως ε, ότι η συνένεση, η συγκατάθεση είναι μία μόνο από τις βάσεις της νομιμοποίησης μίας ε, ε, θεμητής επεξεργασίας των δεδομένων. Αν διαβάσετε την οδηγία θα δείτε ότι υπάρχουν έξι διαφορετικές βάσεις νομιμοποίησης, τρεις εκ των οποίων ε, έχουν μεγάλη σημασία σε σχέση με αυτό το θέμα του consent, της συνένεσης. Ε, πρώτον, στενή έννοια της συγκατάθεσης πέραν κάθε αμφιβολίας. Ε, δεύτερον, contract, σύμβαση. επίσης ε, στενή ερμηνεία της έννοιας γιατί χρειάζεται συγκατάθεση αλλά αν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συμβατική σχέση εφαρμόζονται ελαφρώς διαφορετικοί κανόνες ε, που ε, μπορεί και, και τα δύο είναι σημαντικά στο διαδίκτυο και οι δύο βάσεις. Τρίτον, έχουμε το θεμητό συμφέρον ε, και η ισορροπία που πρέπει να βρούμε σε σχέση με τα ατομικά δικαιώματα και την προστασία τους. Άρα υπάρχει opting out, δηλαδή δεν μιλάμε για opting in, ε, μιλάμε για opting out, δηλαδή μπορεί κάποιος να αρνηθεί να συμμετάσχει. Βλέπετε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Τρεις Τρία διαφορετικά είδη συνένεσης. Ε, ε, παραδοσιακή συνένεση, δεύτερον συνένεση στα πλαίσια μία σύμβαση που ε, προσδιορίζει τι είναι θεμητό και τι είναι όχι και τρίτον άρνηση της συνένεσης, opting out. Και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, την περιπλοκότητα του ζητήματος και τις δυσκολίες εφαρμογής. Κατόπιν, purpose specification, ε, δηλαδή για ποιο σκοπό ε, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Ε, αυτό είναι το κλειδί της αναλογικότητας. Εάν δεν λειτουργούν καλά οι δικλείδες ασφαλείας αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ο στόχος, αν δεν αναφέρεται ρητά από αυτούς που χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Και ένα, μια άλλη βασική αρχή είναι η διαφάνεια, γιατί μας επιτρέπει προβλεψιμότητα, ισότιμη μεταχείριση κτλ. Σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα βέβαια η επιδιωκούμενη διαφάνεια είναι ένας δύσκολος στόχος. Τώρα έχουμε και ε, τεχνολογικές ε, ρήτρες διασφάλισης, ε, ε, δηλαδή να προστατεύσουμε σχεδιάζοντας ε, τους ιστοτόπους με τρόπο ώστε να θωρακίζονται τα ατομικά δικαιώματα όταν δημιουργούνται οι ιστότοποι μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή κάποιου μόνο και μόνο μέσα από τον σχεδιασμό της ε, ιστοσελίδας. Ε, τέλος, ε, βάσει της οδηγίας προβλέπονται και διάφορες εξαιρέσεις ε, για τα δημόσια συμφέροντα που για να τα προστατεύσουμε πρέπει να αναλάβουμε ειδικά μέτρα προβλέπεται αυτό υπό κάποιες επιφυλάξεις. Ε, υπάρχουν και εκεί δίκλειες ασφαλείας και πάλι εδώ πρέπει να ξέρουμε ποια μέτρα θα εφαρμόσουμε και ποιες θα είναι αυτές οι δίκλειες ασφαλείας. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι για την προστασία των ατομικών δεδομένων δεν είναι ισοσκελισμένο το υφιστάμενο πλαίσιο γιατί ισχύει μόνο για τον πρώτο πυλώνα. Ε, εσχάτως υπάρχει και μία απόφαση πλαίσιο για τα θέματα τρίτου πυλώνα. Για το δεύτερο πυλώνα όμως δεν έχουμε πλαίσιο και αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τρεις πυλώνες ε, και αυτό είχε αυξανόμενη σημασία στα πλαίσια του διαδικτύου. Υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες τέτοιες ε, ε, υποθέσεις. Επίσης, ε, εταιρικέ σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το βλέπετε αυτό στο διαδίκτυο. Είναι ένα από το χαρακτηριστικό, ένα από τα χαρακτηριστικά που δημιουργούνται προβλήματα ισορροπίας, ασυμβατότητας λόγω της φύσης του υφιστάμενου πλαισίου και των δικλείδων ασφαλείας. Και στις συνθήκες της Λισαβόνας έχουμε ένα νέο κίνητρο να το δούμε οριζόντια το θέμα ε, ούτως ώστε να καλύψουμε τα χάσματα και να ε, εξαλείψουμε αυτές τις ασυμβατότητες ε, που διαπιστώνουμε. Ε, τώρα ε, ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δρομολογήσει μια open reflection σχετικά με την, τον επίκαιρο χαρακτήρα του πλαισίου μέσα από διασκέψεις σε σεμινάρια τα προσεχή ένα-δύο χρόνια θα εξετάσουμε αυτά τα θέματα όχι μόνο σε σχέση με το διαδίκτυο βέβαια αλλά και γενικότερα. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις ε, επ' αυτού για θέματα που είναι επιτάπητος και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, ε, του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και της προστασίας ιδιωτικής ζωής. Δεν έχω χρόνο τώρα να ε, σε λεπτομέρειες, αλλά αν Μιλώντας για την σημασία της εφαρμογής ε, του υφιστάμενου πλαισίου και των ε, υφιστάμενων αξιών το χώρο του διαδικτύου, είναι ταυτόχρονα σημαντικό να επενδύσουμε σε μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν ότι κάθε φορά που υπάρχει παραβίαση αυτών των κανόνων ε, θα στέλνεται ένα σήμα για την παραβίαση, ένα σημαντικό στοιχείο της αναθεωρημένης οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ένα σημαντικό σήμα, ε, ε συγγνώμη, ε, αυτό το ότι αναφέρεται αυτό μέσα στην οδηγία αποτελεί σημαντικό μήνυμα. Δηλαδή, σε μια διάταξη σχετικά με security breach ε, θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής και να υπάρχουν σαφές Φέστατε διατάξει και να μην περιοριστούμε μόνο σε εταιρείε ε, που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, ε, πάροχοι υπηρεσιών, είτε είναι τράπεζες, ε, είτε είναι ε, Ε, τηλεφωνικές εταιρείες ε, και ξέρω ότι ε, το Συμβούλιο δεν υποστηρίζει πλήρως τη θέση του Κοινοβουλίου αλλά πάντως θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις ε, και να δούμε τις Security Breach Notifications και στο δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι ε, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον του διαδικτύου που ανταποκρίνει το λένε και περισσότερο σε real life situations, δηλαδή σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να ε, δούμε τι θα γίνει με το θέμα του ελέγχου κυρίως ως προς τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου ε, και ιδιωτικού τομέα. Ορισμένες φορές χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και μιλώ για την προστασία των ε, πνευματικών ε, δικαιωμάτων, ε, προστασία του, του επιγραμμικού περιεχομένου και η τάση που υπάρχει να σπρώξουμε κάποιους παρόχους να παρακολουθούν το περιεχόμενο στο ίντερνετ. Τώρα, μέσα στην έκθεση του κυρίου Λαμπρινίδη υπάρχει και ε, μία άλλη έννοια που θέλω να σχολιάσω. Είναι ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πολλαπλοί εμπλεκόμενοι φορείς. Ε, ε, δηλαδή, όλοι καλούνται να διαδραματίσουν το σωστό ρόλο για να έχουμε ένα γενικό καλό αποτέλεσμα. Ε, είναι σημαντικό δεν να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να εμένε το διαδίκτυο να ανήκει στην πραγματική ζωή, στο πραγματικό κόσμο, αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι ε, πλησιάζει περισσότερο ο κόσμος. Ε, τι εννοώ, ότι όταν είσαστε στο διαδίκτυο δεν έχει σημασία που είσαστε, η γεωγραφία δεν έχει πλέον σημασία η γεωγραφική τοποθεσία. Οπότε χρειαζόμαστε πρότυπα, χρειαζόμαστε ένα υγιές, ένα ασφαλές ε, περιβάλλον. Ε, γι' αυτό και ε, πρέπει να υπάρξει υποστήριξη για τον χάρτη των δικαιωμάτων και την εκπόνηση κανόνων, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε τι εστί προστασία των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ρυθμιστικές αρχές διερευνούν τη δυνατότητα εκπόνησης παγκοσμίου προτύπων και ελπίζουν να κάνουν ένα άλμα στον τομέα αυτό κατά το τρέχον έτος, τον Νοέμβριο κατά πάσα πιθανότητα. στη Μαδρίτη. Ε, την επόμενη φορά που θα πάω στην Ουάσιγκτον θα δω σε ποιο βαθμό η νέα κυβέρνηση υποστηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που θα μας επιτρέψουν να γεφυρώσουμε τα χάσματα και να καταλήξουμε σε παγκόσμια πρότυπα. Ε, γιατί είναι σημαντικό να δούμε ποια μηνύματα θα περάσει η νέα κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει διγλώση, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ε, ε, η κατάσταση επιδέχεται βελτίωση για τους ε, χρήστες. Πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση ανάμεσα στους ε, νέους και ηλικιωμένους χρήστες και την ευαισθητοποίηση ε, των νέων. Ο πρόεδρος ομάδας του άρθρου 29 πριν από λίγες μέρες έκανε μια ανακοίνωση σε, από κοινού με την ρυθμιστική αρχή της τσεχικής δημοκρατίας. Δεν ξαφνιάζει αυτό κανένα λόγω της τσεχικής προεδρίας. Ε, σχετικά με τις ε, εκστρατείες ε, ευαισθητοποίησης και αναφέρθηκαν διάφορες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις στον τομέα αυτό. Τώρα, αυτό το περιβάλλον που σας έλεγα με τους πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς, το multi-stakeholder environment, έχει ως αποτέλεσμα ότι χρειάζεται και ρύθμιση και αυτορύθμιση. Χρειαζόμαστε το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά υπάρχει και η εφαρμογή του πλαισίου ε, η οποία θα ενισχυθεί από ε, την επίρρωση των αυτορυθμιστικών μηχανισμών. Και τέλος, ε, κάτι άλλο σημαντικό στο οποίο αναφέρεται και ο κ. Λαμπρινίδης στην έκθεσή του είναι η διακυβέρνηση, το governance του διαδικτύου όπως είναι οργανωμένο δεν έχει πολύ αλλάξει από τις πρώτες μέρες του το διαδίκτυο. Ε, αλλά όταν μιλάμε για απόδοση ευθυνών ε, θα πρέπει να ε, περάσουμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση για την απόδοση ευθυνών και όχι να καταλήξουμε σε ένα υπερρυθμισμένο σύστημα, απλά να αναδιοργανωθεί ο τρόπος ε, ε, οργάνωσης, ε, να αναδιοργανωθεί μάλλον το διαδίκτυο, τόσο ώστε να μπορούμε ευκολότερα να αποδίδουμε τις ευθύνες. Σας ευχαριστούμε, εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η συζήτηση μέχρι στιγμής για όλους όσους έχουν βουτήξει σε αυτό το θέμα. Σήμερα νομίζω ότι λένε και περισσότερο συνειδητοποιούν ε, όλοι την σημασία του ζητήματος ε, και άρα ε, πρόκειται για ανησυχίες εκατομμυρίων πολιτών. Ο καθηγητής πρέπει να φύγει σε 20 λεπτά, ο καθηγητής Ροντότα. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις ή σχόλια για αυτά που μας είπε. Αν θέλετε, κάντε τις ερωτήσεις σας τώρα και θα αποχωρήσει σύντομα. Ποιος ε, ζητάει το λόγο, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Θα μας πείτε και το όνομα σας και την οργάνωση που εκπροσωπείτε. Καλημέρα. Λάμπρος Πατσαβελάς ε, είμαι μέλος της αντιπροσωπείας ε, της Ελλάδας στο Eurojust. Σας ευχαριστούμε για την ε, πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση. Υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου για το Κυβερνοέγκλημα του 2002, 28 Δευτέρα του 2002, και χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο ε, ασχολείται με το ίδιο ζήτημα. Το 2008 καταγράψαμε πολλές υποθέσεις κυβερνοεγκλήματος και για τη διευκόλυνση ανταλλαγής των πληροφοριών ε, δικαστικού χαρακτήρα, δηλαδή εκτέλεση πολλών αιτημάτων αμοιβαία αρρωγής και ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Ε, μπορέσαμε να αποφύγουμε διάφορες ε, περιπτώσεις, όπως βλέπω και στην έκθεση σας, ανησυχεί και σας αυτό το θέμα. χρειάζεται όσοι κάνουν τις έρευνες ε, και όσοι είναι από την εισαγγελία να έχουν τα απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη, να γνωρίζουν τις διερευνητικές μεθόδους τόσο ώστε να ε, λύσουν αυτά τα, τις υποθέσεις ε, κυβερνοεγκλήματος. Είναι το πιο σημαντικό Διεθνέ θέμα και δεν εφαρμόζεται ακόμη ε, ομοιόμορφα το πλαίσιο και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα κολλήματα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση το κυβερνοέγκλημα. Δεν υπάρχει συντονισμό συγκεκριμένα και ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών για ε, τις ε, GIT τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες όταν υπάρχει κυρίως σύγκρουση ως προς τη, προς τη δικαιοδοσία. Ε, και έχουμε... Μην ξεχνάτε ότι το Eurojust είναι πιο πολύ δικαστικό δίκτυο και όχι αστυνομικό, αλλά όλοι καλούνται να συνεργαστούν. Το περασμένο Οκτώβριο κάναμε και το πρώτο σεμινάριο στην Αθήνα για το κυβερνοέγκλημα, όπου... Ε, Συμμετείχαν οι βασικοί φορείς ε, από την ε, ε, Ευρώπη, από τη ΣΥΠΑ, από το χώρο της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου. μπορώ να τονίσω κάποια βασικά ζητήματα. Καταπολέμηση τρομοκρατίας μέσα στο διαδίκτυο, νέοι μέθοδοι πρόσληψης, ριζοσπαστικοποίηση, βασικές υποδομές, προβλήματα που προβλεπούν από τα δίκτυα peer-to-peer, ε, το κατά πόσο μπορούν να γίνουν δεκτά τα ηλεκτρονικά τεκμήρια στα δικαστήρια, ε, μέσα στη συστάση του κ. Λαμπρινίτ προς το Συμβούλιο η δεύτερη είναι σημαντική λέει εκεί ότι πρέπει να ε, εντατικοποιήσουμε τον διάλογο ανάμεσα στο, στα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια και στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νομοθέτες. Είναι πολύ βασικό αυτό και πρέπει να ε, δουλέψουμε ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτό το στόχο και είμαστε στη διάθεσή σας. Ε, αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας. Από πλευράς Eurojust υποστηρίζουμε πλήρως ε, την πρωτοβουλία σας ε, σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και ευχαριστώ όλους τον κύριο Λαμπρινίδη για την αφοσίωσή του στον τομέα αυτό και σας διαβεβαιώ ότι ε, θα είμαστε δίπλα σας, ε, να σας βοηθήσουμε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ. Ε, μία ερώτηση. Σε αυτό το σεμινάριο εκεί στην Αθήνα που είπατε, σκεφτήκατε να καλέσετε παραδείγματος χάρη τον επόπτη, τον, Ευρωπαίο επόπτη προστασίας των ατομικών δεδομένων ή όσοι ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό αυτού αυτοί που ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό, παραδείγματο χάρη των εγκλημάτων, ασχολήθηκαν με το θέμα των ατομικών δικαιωμάτων. Α, κοιτάξτε, ε, ήταν επιχειρησιακού χαρακτήρα η ε, επεξεργασία του ζητήματος από πλευράς μας, ε, δηλαδή συγκεκριμένες υποθέσεις, συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα των ατομικών δεδομένων, αλλά φυσικά Θέλουμε να έχουμε πάντοτε και αυτό ε, το θέμα κατά νου, δηλαδή την προστασία των ατομικών δεδομένων, αλλά απλώ δεν μα απασχόλησε τότε στην Αθήνα. Uh, uh, Για το θέμα της ε, ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και της ανάμειξης του Eurojust. Αλλάξαμε λίγο την... Ε, το πρίσμα γιατί η σχετική σύμβαση ήταν μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, στην οποία ήταν συμβαλόμενα μέρη και πολλές μη ευρωπαϊκές χώρες ε, έχει κυρωθεί από πολλές χώρες η Σύμβαση Προστασίας των Δεδομένων του 1981 ήταν επίσης ανοιχτή σύμβαση για να κυρωθεί και αυτή από μη ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα το Συμβούλιο της Ευρώπης πρόσφατα ε, επεσήμανε αυτή την ιδιότητα αυτής της σύμβασης. Και εγώ θα ήμουν πιο καθυσυχασμένος εάν οι προσπάθειες ε, του ηλεκτρονικού εγκλήματος πήγαιναν χέρι-χέρι με την προστασία των δεδομένων και αντιμετωπίζονταν ως πακέτο. Οπότε, ο ενθουσιασμός που βλέπουμε σε αρκετές χώρες για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και αναφέρατε πως υπάρχουν κάποια ζητήματα μη εφαρμογής. Ο ενθουσιασμός λοιπόν που δείχνουν κάποιες χώρες πρέπει να μας οδηγήσει στο να οδηγηθούμε σε ένα πακέτο για να γίνουν έτσι ακόμη πολύ πιο ισχυρές αυτές οι και νόμιμες οι προσπάθειες αυτές. Σας ευχαριστώ κύριε Σάντσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Σταύρο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις τοποθετήσεις τους και θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις ε, για δύο συγκεκριμένες χρήσεις του ίντερνετ. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας και η προτάσεις σας. Πρώτον, η ηλεκτρονική ψηφοφορία χρησιμοποιείται όλο ένα και περισσότερο στις εκλογικές διαδικασίες ορισμένων χωρών. Υπάρχει περίπτωση εκλογικής νοθείας. Μπορεί αυτό το σύστημα να χρησιμοποιηθεί ε, ε, για τους ε, μετανάστες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ευρωεκλογέ σε λίγο καιρό και πολλοί Ευρωπαίοι δεν μένουν στη χώρα τους. Λοιπόν, τι χρειάζεται ώστε η ψήφος να μην χωρεί νοθείας. Επίσης, προστασία των ανηλίκων. Ο Σταύρος έθεσε ε, ορισμένες ε, ε, οδούς που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι. Εσύ λες στην έκθεσή σου, Σταύρο, ότι, θα, ότι ενθαρρύνεις τους κατασκευαστές ε, κομπιούτερ να εγκαθιστούν προστατευτικά software. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Ευχαριστώ. Καλώς όρισα στην αρχή τον ε, Αλεξάνδρ Άλβαρο και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Πάπα, ο οποίος το ΕΛΚ και να τον ευχαριστήσω και αυτόν για τις βελτιώσεις ε, που έκανε στην έκθεση. Ε, you speak now about cybercrime. I have... Μιλήσατε για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Βεβαίως οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβάνει το να μοιραστεί κάποιος τα προσωπικά του δεδομένα, περιέχει τον κίνδυνο κλοπής της ταυτότητας και το θέμα είναι ποια είναι η θέση σας για το να συμβουλεύουμε τους ε, χρήστες διαδικτύου να έχουν πολλαπλές ταυτότητες για να αποτραπεί η ε, κλοπή ταυτότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση για αυτό το πάνελ, γιατί θα ακολουθήσει και άλλο πάνελ, ας α, ε, ακούσουμε τους ε, ομιλητές μας. Μπορείτε να απαντήσετε και να κάνετε και τις ε, τελευταίες σας παρατηρήσεις. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ροντότα. Το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι ένα ιδιαίτερα αντιμαχόμενο θέμα Υπάρχουν τεχνολογικές ε, πλευρές που αφορούν στην ασφάλεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για να αποφεύγουμε τις νοθείες και ε, περιορίζομαι στο να, λέω, στο να αναφέρω αυτό το πρόβλημα. Τώρα χώρες όπως η Βραζιλία μαζικά προσέφυγαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία αυξάνοντας ε, και την ποιότητα της συμμετοχής ε, διότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία υπάρχουν πολλές ε, μελέτες ιδιαίτερα αντιφατικές μεταξύ τους είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο εγώ θα ξεχώριζα λοιπόν το θέμα της μυστικότητας της ανωνυμίας, της ψηφοφορίας κτλ που είναι πολύ σημαντικό και που κάποιοι είχαν υποτιμήσει κάποια στιγμή λέγοντας εντάξει άσε ψηφίζει ο κόσμος από το σπίτι του με τον υπολογιστή του και μίλησε μάλιστα και για family vote, δηλαδή η οικογένεια ως ε, κοινότητα δεν πρέπει να μετακινείται για να πάει στο εκλογικό κέντρο ε, διότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικής ε, ψηφοφορίας στο εκλογικό κέντρο και η ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία από το σπίτι. Υπάρχει λοιπόν μία κοινή συζήτηση που γίνεται στην οικογένεια και βελτιώνει έτσι και την ποιότητα της συμμετοχής. Λοιπόν εγώ έρχομαι από μία χώρα, την Ιταλία, όπου ε, από μία περιοχή από μια περιοχή όπου η έννοια οικογένεια είναι πολύ διαφορετική. Ξέρετε, η φαμίλια μαφιόζα, οι οικογένειε στη μαφία, οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μεγάλα ρίσκα όταν η οικογένεια δηλαδή αποφασίζει τι θα ψηφίζει. Και η, η είσοδος της ηλεκτρονικής ε, τεχνολογίας κατά τη φάση της ψήφου μπορεί να δημιουργήσει και μία προ πληπτική πρόσβαση στην πληροφορία. Δηλαδή άμα μπω πούμε στην ηλεκτρονική δυναμική της πολιτικής ε, για να ψηφίσω τότε διαπιστώνουμε όπως έγινε και στη Βραζιλία ότι δεν χρησιμοποιεί ο εκλογέας την ηλεκτρονική μόνο για να ψηφίσει αλλά χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να ενημερωθεί κιόλας. Είναι ένα θέμα λοιπόν ε, με πολλές πολλές σημαντικές πτυχές. Δεύτερη γρήγορη θεώρηση. Το θέμα των ανήλικων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι μία υποχρέωση εντό εισαγωγικών του να πρικοδοτήσουμε με διατάξεις όλα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ε, για να προστατεύσουμε τους ανηλίκους είναι πολύ σημαντικά. Λέμε σήμερα ότι για να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι χρειάζεται μια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πιστοποίηση. Αυτό γιατί γίνεται. Για να εγγυθούμε την φυσική υγεία του ανήλικου. Ε, να μην τραυματιστεί, να μην πνιγεί κτλ. Ε, είναι φανερό ότι και αυτές οι τεχνολογίες ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και από αυτήν την πλευρά. Δηλαδή ε, δεν μου φαίνεται ότι θα προκαλούσαν και ιδιαίτερες υπερβολικές δαπάνες επιπλέον από τους παραγωγούς άμα βάλουν και αυτό το προφίλ ασφάλειας. Τώρα το λεπτό σημείο είναι η χρήση της προστασίας των ανηλίκων ε, για κρισία. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα και το επισημένο απλώς. Πολύ πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο στις Ηνωμένε Πολιτείες αποφάσισε για το Child, για το Child Online Protection Act ε, αναζητώντας μία ισορροπία που να μην αμφισβητεί το δικαίωμα του free speech, του ελεύθερου λόγου. Thank you very much, ο Πίτερ Χιούστινγκς. τέλος θα ήθελα να σχολιάσω την κλοπή της ταυτότητας. Το θέμα που ετέθη. Πρέπει να τονίσουμε πως η πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό είναι να διασφαλίσουμε πως οι υπάρχοντες κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μέσο για να υπάρχει σωστή επεξεργασία και λογοδοσία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μπορεί κάποιος με πολλαπλές ταυτότητες στο διαδίκτυο σε αθώα περιβάλλοντα, μπορεί αυτό να είναι μια καλή προσέγγιση Και αυτός είναι ένας τρόπος ε, με τον οποίο μπορούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους οι ενημερωμένοι χρήστες. Εάν όμως έχουμε πολλαπλές αυτοτές π.χ. στην παροχή υγείας, θα έχουμε δραματική μείωση της ποιότητας, θα έχουμε σύγχυση, οπότε δεν θα πρέπει αυτό να είναι έτοιμη απάντηση. Ε, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τονίζουμε την ανάγκη αυστηρής ταυτοποίησης μόνο σε περιπτώσεις εκείνες όπου πραγματικά μετράει η ταυτότητα. Και τονίζουμε την χρήση ε, πραγματικών μέσων ταυτοποίησης όπως ε, διαβατήρια, ηλεκτρονικές ταυτότητες και τονίζουμε την σημασία τους. Απαιτούνται πραγματικά πολύ στιβαρά περιβάλλοντα και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι το τονίζουμε αυτό με ένα συγκεκριμένο σκοπό και μετά επαφίεται σε άλλους χρήστες να βρουν τις συνέπειες. Ε, δηλαδή τι εννοώ, τονίζουμε τα ηλεκτρονικά διαβατήρια γιατί είναι απαραίτητο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κάτι τέτοιο και μετά λέμε εντάξει θα χρησιμοποιηθεί και για άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς σκοπούς. Και έχουμε μπει μετά σε μια κατηφόρα, διολυσθένουμε. Εάν χρησιμοποιήσουμε βιομετρικά στοιχεία για να γίνει ακόμη πιο ασφαλής η ταυτοποίηση στο διαδίκτυο και μετά δεν υπάρχουν διασφαλίσεις για να αποφευχθεί η κλοπή της ταυτότητας, τότε υπονομεύουμε την, την ίδια μας την προσέγγιση. Οπότε αυτό είναι ταυτόχρονα και απαραίτητο και εξαιρετικά περίπλοκο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε συνολικά και να εφαρμόσουμε ε, τα διαφορετικά μέτρα και μετά στο πλαίσιο να είμαστε πολύ αυστηροί. Βέβαια υπάρχουν αυστηρά περιβάλλοντα ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. οι πληροφορίες πιστοτικής κάρτας αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα και το τεχνολογικό ε, περιβάλλον. Π.χ. η διασφάλιση της ιδιωτικότητας ε, από τον σχεδιασμό ήδη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρέπει να επενδύσουμε και σε πράγματα όπως ε, σφραγίδες που δίνουν κάποια λογική ασφάλεια για την ασφάλεια αυτών των περιβαλλόντων και εκεί πέρα πρέπει να σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στα χρόνια που έρχονται. για διάφορους σκοπούς βεβαίως οι πολλαπλές ταυτότητες έχουν νόημα πήγε στο facebook αυτό είναι ε, λογικό καλό είναι να μην είναι κανείς πολύ συγκεκριμένος αλλά αυτό είναι ένας μάλλον πρωτόγονος τρόπος να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας σας ευχαριστούμε Τελειώνει εδώ ο πρώτος γύρος. Ε, επειδή φεύγετε θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, το ερώτημα ήταν για τον κύριο Χάστινγκς. Αυτό. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Μάλιστα, περνάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Να ζητήσω λοιπόν από τον Γκάς Χουσέιν, τον Τζιμ Κίλου και τον Στιβ Πίερς να έρθουν εδώ. Ε, κύριος καθηγητής πρέπει να φύγει. Εσείς κύριε Χιούστινγκς, αν θέλετε να μείνετε, αν θέλετε μπορείτε να μείνετε. Yes me too long. Unbearable. Thanks. I will stay, stay for a while and then Excellent. Okay, okay. Now let me get this chance as the panels are changing. Λοιπόν, ε, καθώς έρχονται οι άλλοι συνομιλητές μας, να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους, συγκεκριμένα την Ειρήνα Βασιλείου στη γραμματεία της Επιτροπής Λίμπε και την ε, κυρία Στεργιάδη, την βοηθό μου, που τα οργάνωσαν όλα αυτά, και για ολόκληρο, ολόκληρο το έργο του για όλη τη δουλειά. I no, no, We'll stay. No, no, thanks a lot. Appreciate it. Okay, apologies for this. Uh, Ωραία, με συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή. Περνάμε λοιπόν στις ευκαιρίε και κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου. Τα εισαγωγικά μου σχόλια νομίζω έθιξαν αυτό το ζήτημα, όπως και κάποια σχόλια των κυρίων Ροντοτά και Χιούστινγκς. Εδώ όμως έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες ε, γνωστούς ε, στον τομέα αυτών, ε, τους οποίους χαίρομαι που καλωσορίζω, τον δόκτορα Γκάς Χουσέιν της Privacy International και επισκέπτη καθηγητή στο London School of Economics, τον Jim Keelock της ομάδας Open Rights και τον Steve Pierce από το Πανεπιστήμιο του Essex που όπως σας είπα ήταν υπεύθυνο για μια έκθεση της Κομισιόν για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδικτύο και την χάρτα δικαιωμάτων του διαδικτύου. Νομίζω ήσασταν εδώ πέρα, ακούσατε το πρώτο μέρος της συζήτησης, οπότε αμέσως θα δώσω τον λόγο στον Δ. Χωσέιν και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε, λέει ο κύριος καθηγητής. Χαίρομαι που ξανά έρχομαι εδώ πέρα. Είναι ενδιαφέρουσε εξελίξει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ουάσιγκτον για κάποιες συναντήσεις και φαίνεται εκεί η αλλαγή της ατμόσφαιρας. Έχει φύγει η κυβέρνηση Μπού, οπότε η ιδέα είναι. Φαίνεται πως εξαρμίζεται, αν θέλετε, η ιδέα πως... Ε, οι ΙΠΑ θα ακολουθούν τι πολιτικές στον πλανήτη. Γιατί ήμουν σε μια συνάντηση όπου ακούστηκε πως ε, οι ΙΠΑ πρέπει να διερευνήσουν το τι θα γίνει με την πολιτική διατήρηση δεδομένων των τηλεπικοινωνιών και θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί το κάνει η Ευρώπη. Δηλαδή πώς φτάσαμε εκεί. Ξεκίνησε η ιδέα στη ΣΥΠΑ, προχώρησε εδώ πέρα και ξαναπήγε στη ΣΥΠΑ. Είναι μια τάση που βλέπουμε στη διαμόρφωση πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνάδελφοί μου και εγώ περάσαμε δύο μήνες ε, ταξιδεύοντας στην Ασία και την Αφρική το καλοκαίρι που μας πέρασε και πάλι το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Συναντηθήκαμε με κυβερνήσεις, ε, αξιωματούχους, ε, κοινωνία των πολιτών, εμπειρογνώμονες και ήταν σαν να ακολουθούσαμε αν θέλετε, τα συντρίμια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όταν ήμασταν στις Φιλιππίνες μας είπαν να πρέπει να κυρώσουμε τη σύμβαση του εγκλήματος του ηλεκτρονικού γιατί μας ε, πιέζει η Ευρώπη». Δεν είχαν ιδέα τι γράφει αυτή η σύμβαση. Ακολουθούσαν κάποιες γελίες πολιτικές. Ε, μιλούσαν για πολιτικές διατήρησης δεδομένων. Και επαναλάμβαναν πως πρέπει να το κάνουμε γιατί το κάνει η Ευρώπη. Ποιος είναι λοιπόν τώρα κακός επιμπούς ε, ήταν η ΙΠΑ. Ε, έγιναν εκλογές, ήρθε άλλη κυβέρνηση τώρα, αλλά η Ευρώπη δεν έχει αλλάξει. Και η Ευρώπη εξακολουθεί να δίνει τώρα το κακό παράδειγμα. Φταίει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, ναι, συχνά ναι, λυπάμαι που το λέω. Στην Αφρική όταν ήμουν μιλούσα στον Υπουργό Μετανάστευσης Κυβέρνησης του Τζιμπουτί και αυτός ε, ήθελε να εφαρμόσει βεβαίως τα δακτυλικά αποτυπώματα για όλο τον πληθυσμό του Τζιμπουτί φεύγοντας τον ρώτησα συγγνώμη με τι λεφτά θα το πληρώσετε αυτά και γελούσε λέει ε, κοιτάξτε μας πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα ε, περίμενα να το χρηματοδοτεί κάτι, κάποιος τσίπα αλλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως σας είπα και στην Κυργυζία ήμασταν πρόσφατα όπου η κυβέρνηση είχε κάποιες αμφιβολίες για το εάν θα έπρεπε να ακολουθήσει ρωσικά συστήματα ε, για την επιτήρηση των επικοινωνιών της, ρωσικά ή ευρωπαϊκά. Και για να είναι σίγουροι έκαναν και τα δύο. Και ήρθαν ε, σε επαφή μαζί μας συνάλφοι από το Πακιστάν το Νοέμβριο, μας είπαν πως φέρνει η κυβέρνηση ένα νέο νομοσχέδιο σχετικό, μου πάνε να το αναλύσουμε και ο νόμος λέει πως ακολουθούμε το παράδειγμα της Ευρώπης ε, αυτό το οποίο μας ζητάει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν διαβάσετε όμως την πολιτική είναι χάλι, μαύρο. Θα βλάψει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, την πρόσβαση ε, στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρουν. Αυτά ξέρουν, αυτά κάνουν. Ε, λένε η κυβέρνηση πως ε, η Ευρώπη τα κάνει αυτά, έχει αυτές τις εξουσίες επιτήρησης και μάλιστα το ηρωνικό είναι πως ε, η σχετική σύμβαση δεν προβλέπει τίποτα για τη διατήρηση δεδομένων. Αυτοί μάλιστα έχουν πάει σε μικρότερη περίοδο διατήρησης δεδομένων από ό,τι ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 9 μέρες, αν και βεβαίως εντάξει, η περίοδος διατήρησης μπορεί να αλλάξει όποτε το κρίνει ο υπουργό. Και λένε επίσης, κοιτάξτε, ακολουθούμε την Ευρώπη, ποινικοποιούμε αυτές τις δραστηριότητες, ε, π.χ. θα τιμωρείται με θάνατο η ηλεκτρονική τρομοκρατία. Αυτό είναι το λαμπρό παράδειγμα που δίνει η Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο. Και όμω πηγαίνουν σε όλε αυτέ τι πρωτεύουσε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και λένε αν δεν περάσετε αυτή τη σύμβαση για την τη τρομοκρατία θα γίνει χαμό. Αλλά όπω ε, σωστά είπε ο Πίτερ Χάστινγκ, γιατί δεν προωθούν και την οδηγία προστασία των δεδομένων. Γιατί δεν ε, προωθούμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε όλο τον κόσμο και μόνο με το ηλεκτρονικό έγκλημα ασχολούμαστε. Οπότε υποτίθεται ότι θα ήταν φωτεινό φάρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση και ανταυτού ε, δίνει το κακό παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια, παρά τι προσπάθειε αρκετών εδώ μέσα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πολιτική διατήρηση δεδομένων και γιατί αλλιώς λέγανε θα γίνει χαμός, οπότε πρέπει να τυποποιηθεί η πολιτική διατήρηση δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση. Και τώρα το σπρώχνει αυτό και η Βρετανική Προεδρία, είχε τότε σπρώξει η Βρετανική Προεδρία. Τώρα πάμε πολύ μακρύτερα. Προτείνουν όλοι οι πάροχοι να αναγκαστούν να εγκαταστήσουν μαύρα κουτιά που θα παρακολουθούν όλη την κίνηση όλων των χρηστών και μετά να πάρουν τα δεδομένα όλα αυτά. Όχι μόνο ποιο στέλνει email, ποιο μιλάει στο Skype, ποιο κάνει chat με ποιον, ποιο έχει φίλου ποιου στο Facebook. Να τα πάρουν όλα αυτά τα δεδομένα οι πάροχοι, να τα στείλουν σε μια κεντρική βάση δεδομένων που θα την βλέπουν μετά όλες οι αστυνομίες του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Αυτό είναι το επόμενο βήμα της διατήρησης των δεδομένων. Και περιέργως πως αυτό προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση Bush με το σκάνδαλο τότε της NSA, αλλά ήταν σκάνδαλο πραγματικά, ζήτησαν να παραπεμφθεί ο πρόεδρος. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και όπως έκαναν και με τη διατήρηση δεδομένων η κυβέρνηση θα πει μα για να είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά. Θα, γίνουν, θα έρθουν λοιπόν στο Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο, θα πούνε πως αν δεν γίνει αυτό θα καταστραφεί ο κόσμος. Και τι θα γίνει, κάθε άλλη χώρα στον κόσμο θα κοιτάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πει αυτό γίνεται στην Ευρώπη, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Πρέπει λοιπόν να σπάσει αυτός ο φαύλο κύκλο γι' αυτό χάρηκα που διάβασα αυτή την έκθεση. Πραγματικά η έκθεση αυτή είναι μια ευκαιρία να αλλάξει το, το ρεύμα, η ροή των πραγμάτων. Είμαι αισιόδοξο γιατί τονίζει τα δύσκολα ζητήματα. Δεν είναι μια γενική δήλωση με τι καλέ ιδέε προστασία των πολιτικών ελευθεριών στο διαδίκτυο. Πραγματικά τα δύσκολα ζητήματα. Απαγόρευση δημιουργία προφίλ. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι γίνεται. Δεν, για τον βαθμό δημιουργία προφίλ που μιλάμε, είτε πρέπει να τα απαγορεύσουμε, είτε τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση. Εδώ μιλάμε για ένα έγγραφο πραγματικά που εδώ και πολύ καιρό είναι το πρώτο που μιλάει για τη συνένεση όχι ως κάτι το υποχρεωτικό για την εκμετάλλευση δεδομένων, αλλά ένα θέμα που αφορά τις σχέσεις εξουσίας. Έχουμε καιρό να δούμε τέτοια σκέψη. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που είδα το πώς θα τα ζητήματα, Ψηφιακή ταυτότητα που ελπίζω να μας οδηγήσει στη δημιουργία μιας ψηφιακής αξιοπρέπειας. Επίσης αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών από τρίτα μέρη ουσιαστικά πράγματα και τα ξέρει ο κλάδος. Όλοι ξέρουν πως είναι ουσιαστικό αυτό γιατί υπάρχει αυτός, αυτό το οποίο λέμε cloud computing, ότι θα πάμε προς το να γίνονται όλες οι εργασίες στο διαδίκτυο. Αλλά αν δεν περιοριστούν αυτές οι εξουσίες πρόσβασης των αστυνομιών, δεν θα συμβεί αυτό ποτέ. Κανείς δεν θα έχει εμπιστοσύνη στο δίκτυο. Οπότε έχετε πραγματικά ένα όραμα και είναι τιμή που είμαι εδώ και, να, και το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ πέρα. Μιλάτε για το πώς πρέπει να εμποδίσουμε τη συστηματική παρακολούθηση όλων των ε, δραστηριοτήτων. Δεν ξέρω αν μιλάτε και για την διατήρηση δεδομένων, γιατί αν ε, το συμπεριλαμβάνει είναι πολλά υποσχόμενο, εάν όχι όμως δεν έχουμε λύσει τίποτα. Κατά κάποιον τρόπο η διατήρηση των δεδομένων ε, έχει μεταμορφώσει τη σχετική νομοθεσία λέγοντας πώς η απλή συλλογή των δεδομένων δεν είναι επέμβαση στην ε, προσωπική ζωή του ατόμου. Τεράστια αλλαγή νοοτροπία. και αν δεν το αλλάξουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τίποτα. Δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις ε, τοπικές αυτοδιοικήσεις, αστυνομίες, τον οποιονδήποτε θέλει. Και εμείς θα λέμε πω δεν είναι η επεξεργασία, είναι η συλλογή ήδη εισβολή στην ιδιωτική ζωή. Οπότε είμαστε σε μια πολλά υποσχόμενη στιγμή αυτή τη στιγμή. Επίσης λυπούμε για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε την κυβέρνηση Μπούσος το παράδειγμα ανά τον πλανήτη. Έχουμε μια ευκαιρία να τα αλλάξουμε. Πότε θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Μπούσος έφυγε λόγω εκλογών. Έχουμε εκλογές σε κράτη-μέλη, έχουμε εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά υπάρχει μία συγκεκριμένη στιγμή που θα έρθουν νέες ιδέες και θα υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα πριν και το μετά. Για να τελειώσω λοιπόν, έχουμε μια πολύ συναρπαστική ευκαιρία αυτή τη στιγμή, ευκαιρία που δεν έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Περνάμε στον Jim Killock τώρα, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του, του οργανισμού της ομάδας Open Rights. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Okay, thank you. Um, so, Ουσιαστικά εγώ θα σας μιλήσω για τις ανησυχίες που έχουμε στην ομάδα μας, στην Open Rights, σχετικά με ε, τις επιπτώσεις ε, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ε, καθώς και τις επιπτώσεις των δράσεων των εθνικών κυβερνήσεων και συγκεκριμένα τις δράσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί εμείς ε, σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιούμαστε ως επιτοπλίστων. νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για τις θετικές πτυχές. Θεωρούμε εμείς πως ε, είναι πολύ θετικές οι ευκαιρίες που μας προσφέρει το διαδίκτυο, δηλαδή η πολιτική συμμετοχή, δημοκρατική συμμετοχή και αυξημένη διαφάνεια. Ε, ε, η κοινωνία των πολιτών μετεξελίσσεται ραγδαία, αλλά αυτό το θέμα είναι, παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής διαβλέπουμε κινδύνους ε, παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και αυτό σχετίζεται με το νομικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε και ε, την ε, αυξημένη προσοχή που πρέπει να δείξουμε σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι ψηφιακές πληροφορίες αντιγράφονται εύκολα, αποθηκεύονται εύκολα, πιο φτηνά και ε, μπορούμε να τις, ε, ε, και οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία μπορούν εύκολα να τις αναλύσουν αυτές τις αποθηκευμένες πληροφορίες και αυτό εγκυμονεί διάφορους κινδύνους. Ε, και μιλάμε για διάφορα εγκλήματα που συμβαίνουν στον ε, κυβερνοχώρο, Παραδείγματο χάρη παραποίηση ταυτότητας ε, που σχετίζονται με τη χρήση των δεδομένων, παραβίαση της ατομικής ζωής, κακοδικίε κτλ. Και σε σχέση με τον τρόπο που εκδικάζονται οι υποθέσεις, υπτίθεται το θέμα της συλλογή των δεδομένων και της ανταλλαγής ανάμεσα στις εταιρείε, αλλά υπάρχει και το θέμα της ανθρώπινης αξιοπρόπειας. Δηλαδή όλοι κρινόμαστε από αυτά που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ε, κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες λόγω ε, ε, μιας παρελθούσας συγκυρίας. Δεν έχει καμία σχέση με τις τωρινές ανάγκες του ατόμου. Έχουμε και μια δημοφιλή σειρά στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου γελιοποιούμε αυτή την κατάσταση, τη διακομωδούμε και λέει ο υπολογιστής όχι κάθε φορά που κάποιος υποβάλλει αίτημα για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας. Αυτό είναι σοβαρή ε, ανησυχία. Ε, έχουμε το data mining, ε, έχουμε τους τη χρήση των δεδομένων κατά των μακροχρόνια ανέργων. Ε, δηλαδή ε, μπορεί να υπάρξει σαφή σε διακριτική μεταχείριση και είναι δυσδιάκριτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη χρήση των δεδομένων και, στην, ε, τη διακριτική μεταχείριση των ατόμων σε σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές ε, και τη δράση τους για αυτές τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες, ε, συχνά ε, έχουν την τη τάση οι άρχες να χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη την Oyster Card για τα ταξίδια το που κάνουμε, για τις κρατήσεις που κάνουμε για εισιτήρια και χρησιμοποιούνται τα στοιχεία για λόγους διατήρησης δεδομένων, ε, πέραν δηλαδή από τον αρχικό σκοπό της υπηρεσίας, οπότε παραβιάζεται η ατομική ε, ζωή. Ε, τώρα το ίδιο το σύστημα, στο ίδιο το σύστημα δεν διευκρινίζεται γιατί υπάρχει αυτή η λειτουργία, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα γιατί έχει προβλεφθεί αυτή η λειτουργία. Ε, Παραδείγματο χάρη στην αστυνομία έγιναν δεκτά 400 αιτήματα για ε, Oyster Cards για εξάμηνη περίοδο Δηλαδή ε, από τον Αύγουστο του 2004 μέχρι τον Μάρτιο του 2006 ζητήθηκαν δεδομένα και η αστυνομία ε, μπορεί να κάνει την ε, παρακολούθηση αυτή χωρίς να υπάρχει η έγκριση κοινοβουλευτική. Αν το σκεφτείτε καλά, τα δεδομένα για τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών υπερβαίνουν τις δυνατότητες παρακολούθησης ακόμη και της μυστικής αστυνομίας ε, ε, δηλαδή που λειτουργούσε πριν από 30 χρόνια σε κράτη όπου φυσικά η τεχνολογία δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη εκείνη την εποχή η πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία τα, από τις αρχές επιβολής νόμου πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει επαρκή εποπτεία αυτών των δραστηριοτήτων, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και μελλοντικά προγράμματα όπως ε, το Μητρό των ε, Ταυτοτήτων ε, και το ΣΥΣ, το Σύστημα Πληροφοριών του Σέγγεν, μας ανησυχεί γιατί υπάρχουν ηθικές επιπτώσεις για την ανταλλαγή των πληροφοριών και την, το λεπτομερές profiling της ζωής κάποιων ανθρώπων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν επίσης τεχνολογίες ε, για ε, ε, την αυτόματη καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας και ε, υπάρχουν ε, πληροφορίες που διατηρούνται από, ε, για ένα έως πέντε χρόνια χωρίς να υπάρχει συζήτηση και χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική έγκριση. Οπότε είναι πολύ σοβαρή πρόκληση αυτή η σώρευση των ατομικών δεδομένων χωρίς να έχει πληθεί της υπόθεση ο αρμόδιος επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παρακολούθηση και για τον έλεγχο. Πολλές ε, ανησυχίες έχουμε σε σχέση με τις πολιτικές ελευθερίες ε, ε, πρόσφατα. Αναφέρθηκαν σε οι τεχνικές data mining και υπάρχει και το θέμα της αλογικότητας που πρέπει να, η αρχή πρέπει να τηρείται όταν, στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων. Ε, υπάρχουν ε, σοβαρές απειλές ε, στο στην ψηφιακή μας ύπαρξη, όπως παραδείγματος χάρη παραπέμπει ταυτότητα. όταν υπάρχει απώλεια δεδομένων, ε, αλλά αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Είναι από αποτέλεσμα τεχνολογικών μέτρων και συστημάτων που οδήγησαν σε αυτά τα προβλήματα. Ε, η ασφάλεια των υπολογιστών, παραδείγματο χάρη, γιατί από αυτό εξαρτάται η προστασία της ατομικής ζωής, ε, είναι κάτι που παραμελείται. Υπάρχει το θέμα της κρυπτογράφησης. Λένε κάποιοι ότι ε, ε, δεν λειτουργούν σωστά ε, τα συστήματα, ότι δεν είναι προβλέψιμη η ανθρώπινη συμπεριφορά και ότι σε αυτό οφείλεται αυτός ο κίνδυνος. Τώρα για την ανταλλαγή των δεδομένων, χρειάζονται ασφαλείς ε, βάσεις ε, δεδομένων ε, στις οποίες έχουν πρόσβαση όμως εκατομμύρια χρήση και τεχνικώς πώς αυτό είναι ανέφικτο. Δυστυχώς αυτοί που εκπονούν τη δημόσια πολιτική δεν τον λαμβάνουν αυτό υπόψη και και στις ε, βασικές ε, θέσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπάρχουν ικανοί επιστήμονες ε, στον τομέα της πληροφορικής που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα της κεντροποίησης των δεδομένων σε βάσεις ε, και όσοι αναφέρονται στα ενδεχόμενα προβλήματα ε, παραγωνίζονται και ε, αφήνεται όλη η ευθύνη σε εμπορικούς παρόχους υπηρεσιών. Ε, στην, ε, υπάρχει η σχετική επιτροπή για την ε, κοινωνία της πληροφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί υπέβαλα αυτό ακριβώς το ερώτημα. Αν υπάρχει στη δική τους υπηρεσία ας πούμε ένας επιστήμονας στον τομέα της πληροφορικής και είπαν όχι ακόμα. και είπαν ότι μόλις βρούμε τα λεφτά θα προσλάβουμε κάποιον. Μα είναι απαράδεικτη αυτή η προσέγγιση σε μια περίοδο που επιδιώκουμε την εναρμόνιση των βελτίστων πρακτικών σε, σχέση, σε όλες τις υπηρεσίες πληροφορικής όλων των κρατών μελών. Ε, υπάρχει και ο Ευρωπαίος Επόπτης έτσι, για τα ατομικά δεδομένα που είναι ένα καλό παράδειγμα ε, και... όπως ανέφερε υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές αλλά όχι στα μεγαλύτερα κράτη-μέλη και δεν είναι, ε, ξέρετε, αναδρομικά εύκολο να ε, επιβάλλουμε συνθήκες ασφαλείας σε ένα σύστημα. Πρέπει εξ αρχής να το προβλέψουμε. Ε, υπάρχουν καταγγελίες πάντως από ειδικού στον τομέα της πληροφορικής σχετικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας στα κυβερνητικά προγράμματα ε, και υπάρχει και το κόστος ε, των ε, συστημάτων. Ξέρετε, εύκολα μπορεί κάποιος να κόψει το κονδύλι σχετικά με την ασφάλεια. αλλά όμως σε αυτό βασίζεται η προστασία της ατομικής μας ε, ζωής, οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια ως έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη δράση των κυβερνήσεων. για την υποκλοπή των δεδομένων ε, από τις ε, κυβερνήσεις επίσης ε, υπάρχουν πολλές ανησυχίες από τις ομάδες προστασίας των πολιτικών ελευθεριών. Οι εταιρείε μας, παραδείγματος χάρη για πολύ μεγάλη περίοδο, αποθηκεύουν δεδομένα ε, κάτι που δεν προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, απλώς προβλέπεται στη δική μας νομοθεσία και το εξάγουμε το σύστημα. Αυτή η διατήρηση δεδομένου μας λένε είναι απαραίτητη για να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα και την τρομοκρατία, αλλά δεν υπάρχουν τεκμήρια και τα δεδομένα ε, χρησιμοποιούνται για πληθώρα άλλων στόχων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, δεν υπάρχει δικαστική εποπτεία και, ε, δεν, ε, και υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που μας οδηγούν σε γελίες καταστάσεις, δηλαδή τοπικά νομικά συμβούλια ζητούν, παραδείγματο χάρη, να ε, ελέγξει κάποιο αν είναι, μπορεί να είναι επιλέξιμα κάποια παιδιά για να μπουν σε συγκεκριμένα σχολεία, παραδείγματο χάρη. Ε, τώρα για τις τηλεπικοινωνίες και τα σχετικά δεδομένα, για, ε, για τα email, για τα SMS, παραδείγματος χάρη, ε, διευρύνονται αδικαιολόγητα οι εξουσίες ε, της ε, κυβέρνησης για τη διατήρηση των δομένων. Κανείς δεν έπαιρνε 200 γράμματα την ημέρα στο, στο παρελθόν και εν περιπτώσει δεν μέσα δεν επικοινωνούσαμε διαρκώς με τους φίλους μας στο ίντερνετ, δεν κουτσομπολεύαμε στο βαθμό που κάνουμε τώρα διαδικτυακά. Αλλά για όλα αυτά τώρα υπάρχουν ε, ε, ηλεκτρονικά αρχεία ε, που διατηρούνται σε ή μη κρατικά φόρα. Αυτή είναι ημικρατικά κρατικα φορα αυτη παραβίαση της ατομικής μας ζωής, κυρίως όταν μιλάμε για αυτά τα ίχνη, τα footprints, ε, τα οποία όμως δεν γνωρίζει το κοινό. Ε, και αυτό μπορεί να τροποποιήσει αρνητικά την ε, συμπεριφορά μας. Ε, Παραδείγματο χάρη μια ριζοσπαστική Ισλαμική ε, ιστοσελίδα. Ε, αν τη συγκρίνουμε με μια εθνικιστική ιστοσελίδα, Είναι κακό να επισκεφτεί κάποιο ε, τι σελίδε. Ε, πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση σε περίπτωση κρίση όπω στη Βόρεια Ιρλανδία ε, για ομάδε αμφισβητούμενη νομιμότητα. Εκεί πέρα πώ μπορεί κάποιο να αποφασίσει αν υπάρχει παραβίαση ή όχι. Ε, τώρα στραφώ προς τον ιδιωτικό τομέα εκεί. Ασκούνται διαφορετικές επιώσεις ε, και ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη γιατί υπάρχει και το θέμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά τη διατήρηση των δεδομένων. Εμείς ένας καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη υπηρεσία. Οπότε αλλά επίσης ε, ε, ε, εξεγείρονται αν θέλετε κάποιοι καταναλωτές και αλλάζουν οι πρακτικές κάποιων εταιριών όπως του Facebook παραδείγματο χάρη. Ναι, πρέπει να είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις αλλά πρέπει να αποθηκεύονται τα δεδομένα και να την χάνουν διαφανούς επεξεργασίας και εύκολα να μπορεί να υπάρχει αναδρομικά ανάκληση των ισχύουσων διατάξεων κυρίως ε, στη ΣΥΠΑ όπου μιλάμε για πολύ διαφορετική κειμένη νομοθεσία δηλαδή υπάρχει το, η γνωστή Patriot Act, η νομοθεσία που δίνει ε, τέτοιες αρμοδιότητες ε, στην κυβέρνηση τον είπα για την αποθήκευση και τη διατήρηση των δεδομένων ε, δηλαδή είναι υπέρ του κράτους και όχι υπέρ του ατόμου υπάρχουν και ρυθμιστικά προβλήματα δηλαδή οι χρήστες δεν κάθεται να διαβάσουν τους όρους χρήσης ενός ιστοτόπου δεν δηλαδή κάνοντας ένα κλικ με το ποντίκι ε, ε, ε στο ναι δέχομαι τους όρους, ε, δεν σημαίνει ότι τους έχουν διαβάσει και όλους, πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση για να καταλαβαίνουν οι χρήστες περί όσο επρόκειται. Ε, και να ένα παράδειγμα πώς ακριβώς μπορούμε να είμαστε πιο φιλικοί προς το χρήστη και όχι να μην έχουμε μια απλά νομική προσέγγιση. Ε, και θα χρειαστεί να προωθήσουμε οποιασδήποτε καλές πρακτικές υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, τώρα, ε, για την ενίσχυσή της ιδιωτικής ζωής, το PGP, και διάφορες εταιρείες όπως η Microsoft προβάλλουν τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες μεταβίβασης ατομικών ε, δεδομένων και μπορεί να είναι πολύ χρήσιμε στο μέλλον αυτές οι τεχνολογίες. Αλλά ε, υπάρχει και το θέμα της ε, διαφήμισης. Εδώ εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες γιατί το Internet Advertising Bureau εξέτασε το θέμα του κώδικα διοντολογίας και ένα σύστημα για τα cookies με δυνατότητα opting out για το behavioral advertisement ε, ούτως ώστε επανειλημμένα όταν αλλάζει κάποιος browser ή σβήνει τα cookies ή αλλάζει υπολογιστή να έχει αυτή τη δυνατότητα opting out ε, και για την προστασία των δεδομένων. Μόλις γίνει μια επιλογή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, δεν θα πρέπει να μπορεί να ανακληθεί. Εάν ε, δηλαδή η τεχνολογία δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή την επιλογή θα πρέπει να την διαμορφώσουμε την τεχνολογία ή να τη χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά. Αλλά ας δούμε και τα είδη των δεδομένων που συλλέγονται, είτε μιλάμε για να αποφασίσουμε αν είναι καλύτερο το opting in ή το opting out, για την ε, browsing history παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι το παράθυρο προς την ψυχή σας, λέει πολλά πράγματα για το άτομό σας. Ε, ε, και ορισμένε φορέ γίνεται η επιλογή να διαβάζει ούτως ή άλλως όλα τα δεδομένα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο η βιομηχανία ποια στάση θέλει να τηρήσει, αν ε, θέλει να συμπεριφερθεί σε θελοντική βάση, να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση, δηλαδή όπου υπάρχει επιλογή και γίνονται όλα σε θελοντική βάση ή όχι. Ε, τώρα υπάρχει υπηρεσιών, ε, χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες ε, και μην ξεχνάτε όμως ότι είναι... Μέσα στις ιστοσελίδες ε, υπάρχουν δεδομένα ατομικά ή δημόσια διαθέσιμα, αλλά δεν ε, χρειάζεται, δεν ζητείται συγκατάθεση των αρμοδίων για τους ιστοτόπους ώστε να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση, όχι σε όλες τουλάχιστον ε, και ε, θα πρέπει να προστατεύονται οι καταναλωτές, οι χρήστες δηλαδή των ε, ιστοσελίδων από τις ίδιες τις ιστοσελίδες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ενημέρωση προς τους καταναλωτές ότι μπορεί κάποιος να έρθει και να ελέγξει τα δεδομένα που έχουν ε, ανεβάσει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αλλά αυτή είναι η μία πλευρά ε, και θεωρούμε ότι Ε, δεν ε, υπάρχει σαφής αντίληψη περί του κονσέν της συγκατάθεσης του καταναλωτή όταν μιλάμε για τέτοιες ε, διαφημίσεις και Ελπίζω οι ιστοσελίδες να μεριμνήσουν, ε, οι υπάροχοι δηλαδή να μεριμνήσουν ούτως ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και ε, πραγματικά ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, εμπειρογνώμονες, επιστήμονες στον τομέα της πληροφορικής, μόνο εκείνοι μπορούν να διαφυλάξουν τα δικαιώματα των χρηστών, μόνο έτσι μπορεί να επικρατήσει μεγαλύτερη διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει απόδοση ευθυνών για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και το οικονομικό μοντέλο θα πρέπει να αρχίσει να αντανακλά τους κινδύνους κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη ασφάλειας και η διατήρηση των δεδομένων είναι ένα θέμα που πρέπει να επανεξετάσουμε για να καταλάβουν οι καταναλωτές ε, επιτέλους ότι ουσιαστικά ιδιωτική ζωή δεν έχουν πλέον. Ε, finally, ε, Professor Thank Τέλος, ε, ο καθηγητής ε, Πίερς, ε, ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Έχω την ευκαιρία, είχα και την ευκαιρία νωρίτερα να εκπονήσω μια μελέτη για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της έκθεσης και να κάνω και κάποια επιπρόσθετα σχόλια. Ε, η μελέτη έχει δύο τμήματα. Πρώτον εξετάζει ε, το θέμα του διαδικτυακού ε, χάρτη δικαιωμάτων και μετά ε, ασχολείται με το κυβέρνο έγκλημα. Αλλά υπάρχει και σχέση, ένας δεσμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο τμήματα της έκθεσης ε, και ασχολούμαστε με το θέμα της νομοθεσίας για τα κυβέρνο έγκληματα και πώς αυτό επηρεάζει τα ατομικά δικαιώματα. Και πάλι εδώ είναι αμφίδρομη η διαδικασία. Υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει τα ατομικά δικαιώματα, άτομα για την ιδιωτική ζωή, καταναλωτικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται ποδέ γενικότερα σε χάρτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά υπάρχει και νομοθεσία που ε, καλύπτει το ζήτημα της προστασίας ε, των δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη το δικαίωμα της έκφρασης ή της ελευθεροτυπίας. Υπάρχει αρχικά η ιδέα ενός ε, διαδικτυακού χάρτη δικαιωμάτων και ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με αυτό το θέμα είναι διότι μέσα στην ε, εντολή που είχα ε, στην έκθεση που συνέταξα τίθεται αυτό το ζήτημα αν χρειαζόμαστε ή όχι ένα χάρτη τέτοιων δικαιωμάτων και το βασικό ζήτημα είναι αν αυτό συνιστά προστιθέμενη αξία ως προς την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων ούτως ώστε να είναι πιο να Βάλετε περισσότερη νομοθεσία ή να διευκρινίσουμε πώς ακριβώς θα προστατεύουμε τα ατομικά δικαιώματα στα πλαίσια του διαδικτύου, ε, αυξάνοντας, ε, τον, ανεβάζοντας τον πύχη ή θέτοντας ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την ε, προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Δεν προτείνω να συντάξουμε ένα νέο δεσμευτικό έγγραφο Απλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε πώς τα υφιστάμενα επίπεδα προστασίας μπορούν να εφαρμοστούν στο ε, ίντερνετ και πώς ε, μπορεί να υπάρξει ευρεία συγκατάθεση, ευρεία συνένεση ανάμεσα σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς και ίσως να να προβάλλουμε και αυτό το Bill of Rights ή όποιο είναι το έγγραφο στο οποίο θα καταλήξουμε. Για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση δεν προτείνω... Ε, δεν ε, ε, θεωρώ ότι αυτό είναι το έγγραφο οπωσδήποτε πρέπει να συντάξουμε ή ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Απλά το Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθεί με τις ίδιες τις χρήσεις του διαδικτύου για να αναλυθεί μια πρωτοβουλία και να καταλήξουμε σε κάποιο έγγραφο. Αν η πρωτοβουλία αυτή ε, ξεφύγει από το πλαίσιο της Ένωσης, μπορεί το έγγραφο να διαφέρει από άλλες ε, διεθνείς δεσμεύσεις ε, άλλες συμβάσεις προστασίας των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και άρα θα πρέπει να αναδιατυπώσετε το κείμενο και θα προκύψει ένα νομικό πρόβλημα. Θα υπάρξει μια σύγκρουση δικαίων. και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι ε, να μεριμνήσουμε το ώστε στο διαδίκτυο να μην υπάρχει χαμηλότερη προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Τώρα, πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών ή σε ποιο βαθμό θα εμπλακούν οι εταιρείες. Ε, δηλαδή το Google παραδείγματο χάρη είναι μια εταιρεία ανάμεσα σε άλλες ε, που καλείται να αναλάβει ένα ρόλο στη, για την προστασία δεδομένων αλλά αυτό δεν μπορεί να, δεν μπορεί κάνουμε παραλληλισμό με μια μη κυβερνητική οργάνωση γιατί υπερασπίζονται τα συμφέροντά της υπερασπίζεται τα σφαιροντά ε, η συγκεκριμένη εταιρεία. Ε, το Google λοιπόν ε, και άλλες τέτοιες εταιρείες πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία γιατί αλλιώς δεν θα είναι αποτελεσματική η διαδικασία αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει απλώς να τους δώσουμε μια λευκή επιταγή. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το δούμε αρχικά το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, δεν έχει αναπτυχθεί αυτή η ιδέα για την προστασία των ατομικών δεδομένων ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε γίνει παλιά αυτή η συζήτηση, αν ήταν καλύτερα να γίνει ε, η συζήτηση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ε, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν κάποιοι οργανισμοί του ΟΗΕ για την ελευθερία, για να θυμιστεί θέμα της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας της. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι διδή προσέγγιση και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ακούσαμε, αν ε, πρέπει να αναφερθούμε στα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία, ε, τα δικαιώματα, εγώ τα έβαλα στον κατάλογο ε, γιατί σχετίζονται άμεσα με το διαδίκτυο, αλλά υπάρχει και το αντίθετο επιχείρημα ότι δηλαδή οι δισκογραφικές εταιρείες και όσοι παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο δεν χρειάζεται να αναφερθούν στα ε, πνευματικά δικαιώματα. Μπορούμε να ε, ε, αναφερθούμε και στα εμπορικά δικαιώματα μέσα σε αυτό το χάρτη δικαιωμάτων. Αλλά το βασικό είναι οι καταναλωτέ να προστατεύεται η προστασία τη ελευθερία έκφραση, να προστατεύονται οι χρήστε, να προστατεύονται τα παιδιά κτλ. Για να δούμε τα ζητήματα του εγκλήματο. Υπάρχει η Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για αυτό το θέμα και μέσα σε αυτή το πρωτόκολλο όπου μιλάμε για το ρατσισμό την ξενοφοβία. Και μετά η ίδια η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για την πρόληψη της ε, τρομοκρατίας ε, και τέλος η τελευταία σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών. Όλες αυτές οι συμβάσεις εν μέρη σε μεγάλο ή μικρό βαθμό ασχολούνται και με αυτά τα θέματα τα επιγραμμικά, τα online. Τώρα ε, υπάρχει προστασία μέσα από αυτά τα μέτρα, αλλά ενέχονται και κίνδυνοι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περνάω τώρα σε αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μικρότερο βαθμό τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ε, στα, σε σχέση με αυτά τα μέτρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τι έχουν κάνει λοιπόν. Ε, έχουν εφαρμόσει μέτρα τρίτου πυλώνα μέσα στην ε, κοινοτική νομοθεσία ε, έχουν εφαρμόσει διάφορες διατάξεις από όλες αυτές τις συμβάσεις ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης που προανέφερα. εν μέρη έχουν εφαρμοστεί αυτές οι διατάξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις ε, συμβάσεις αυτών και το πεδίο εφαρμογή των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εν μέρη έχουν εφαρμοστεί οι συμβάσεις ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα μέτρα που πρότεινε μέσα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα εφαρμόζεται σε όλη τη... Ε, τα μέτρα τα κοινοτικά εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ισχύει για όλα τα μέτρα ε, που προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και επίσης υπάρχει και το θέμα της νομολογίας του ΔΕΚ και οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηριών που δίνουν την ερμηνεία κάποιων νομοθετικών διατάξεων και υπάρχει και το θέμα των ε, προσφυγών ε, όπως έγινε παραδείγματος χάρη για την ε, οδηγία διατήρησης δεδομένων προσφυγών για ακύρωση παραδείγματος χάρη Τώρα, το θέμα της ασφάλειας των δικτύων ε, δεν καλύπτει την χρήση του διαδικτύου από τους καταναλωτές ε, γιατί μιλάμε για παράνομη υποκλοπή ε, των δεδομένων. Αυτό προβλέπεται στη σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα αλλά δεν αποτελεί έτσι ακέραιο ε, κοινοτικό μέτρα, μέτρο και επίσης ε, το θέμα της ε, παραποίησης ταυτότητας του phishing επίσης που προβλέπονται σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο κοινοτικών μέτρων. Ε, και έγινε και μια μελέτη σχετικά με το αν πρέπει να υπάρξουν κοινοτικά μέτρα γιατί είναι τόσο διαδεδομένο φαινόμενο και θα πρέπει να δούμε ε, σε ποιο βαθμό ε, η εναρμόνιση της νομοθεσίας σε κοινοτικό επίπεδο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαδραματίσει ρόλο τόσο ώστε να προστατευτούμε αποτελεσματικά κατά αυτών των μέτρων. Θα επανέλθω στην παράνομη υποκλοπή των δεδομένων στη συνέχεια. Τώρα, σεξουαλική εκμετάλλευση κακοποίηση των παιδιών υπάρχει απόφαση πλαίσιο που έχει ευρύτερο ε, πεδίο εφαρμογή σε σχέση με τη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για το κυβερνοέγκλημα. Επίση, παιδική πονογραφία, έχουμε του ορισμού, τι πρέπει να ποινικοποιείται από τα κράτη-μέλη. Είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογή, αλλά έκτοτε προέκυψε και η Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την προστασία των παιδιών, που εν γέννη είναι ευρύτερη από τα μέτρα τα κοινοτικά το θέμα τώρα. Είναι η Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να φτάσει στο επίπεδο τη Σύμβαση ε, του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την προστασία για το παιδιών, γιατί ακόμα λίγα κράτη-μέλη την έχουν προσυχογράψει. Ε, ε, ο Επίτροπος μέχρι το τέλος του μήνα θα κάνει μια πρόταση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ε, ξεχωριστές συστάσεις για το ζήτημα αυτό, για θέματα όπως grooming ή επιγραμμική πρόσβαση σε ιστοτόπους υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ε, είναι απαραίτητο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσουμε τα παιδιά κυρίως από τις ακραίες ε, μορφές εκμετάλλευσης, ε, δηλαδή επαφή με ένα παιδί για σεξουαλική εκμετάλλευση, για κακοποίηση, όπως στην περίπτωση του grooming ή για την παιδική πορνογραφία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει ε, προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είναι μέρος της πρότασής μας. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Οι συστάσεις του κοινωνικού Κοινοβούλιο που εγκρίθηκαν ήδη, είπαμε, σε αυτό το τομέα προτείνουν ε, τα, ε, ε, τα chat rooms των παιδεραστών να ποινικοποιούνται. Το chat room τώρα σε, σε ποιο μέτρο είναι ένας μηχανισμός που, που επιτρέπει την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Δηλαδή αν κάποιος απλώς συζητεί το θέμα και είναι πολύ αμφιλεγόμενη η άποψή του σε σχέση με το να υπάρχει χαμηλότερο ηλικιακό όριο για την, ε, να θεωρηθεί ότι ένας ε, ανήλικος έχει ε, δώσει τη συγκατάθεσή του για μια σεξουαλική πράξη παραδείγματο χάρη, σε, σε ποιο βαθμό ποιο, θα αποφασίσουμε αν πρέπει να ποινικοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε ένα chat room σε κάθε περίπτωση και σε σε, ε, στο να έχει κάποιος και να δια, ε, διαδίδει ε, δεδομένα μάλλον υλικό παιδικής πορνογραφίας, παραδείγματος χάρη. Ε, και είπε κάποιο ότι το πρέπει και σε ψηφιακό επίπεδο και σε πραγματικό επίπεδο να προστατεύονται τα παιδιά, αλλά ξέρετε το υλικό παραδείγματο χάρη, τα κινούμενα σχέδια παιδική πορνογραφία ε, ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί να ταυτιστεί με την ίδια την σεξουαλική κακοποίηση ενό παιδιού στον πραγματικό κόσμο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε το ψηφιακό υλικό, ούτως ή άλλως μεγάλο βαθμό γίνεται η μέσα μέσα στην απόφαση πλαίσιο. Απλά η προτεραιότητα μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι η ουσιαστική προστασία των πραγματικών παιδιών έτσι, κατά της ε, ε, παραγωγής τέτοιου πορνογραφικού υλικού ή της σεξουαλικής τους ε, κακοποίησης. Ε, για το θέμα της ε, τρομοκρατίας, που, στο οποίο αναφέρθηκαν οι και οι συνάδελφοι, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει ήδη απόφαση πλαίσιο που αντιγράφει τα τρία βασικά εγκλήματα της ε, Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 και διευρύνει τις υποχρεώσεις της Ένωσης σε σχέση με αυτή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε και έχουν αντιγράψει τους ορισμούς των εγκλημάτων, αλλά ο ορισμός της τρομοκρατίας, παραδείγματος χάρη, διαφέρει ε, και το θέμα της δικαιοδοσίας διαφέρει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι έχουμε ένα κοινό ορισμό Μιλάμε για πολύ ευρύτερη απαγόρευση. Αυτήν έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι προβληματικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν μιλάμε για την ε, απαγόρευση τη ε, δημόσια παρακίνηση τη τρομοκρατική ενέργεια που δεν έχει καμία σχέση με την ίδια την τρομοκρατική πράξη. Απαγόρευση δηλαδή δημοσίων δηλώσεων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραδείγματο χάρη και αυτό διαφέρει από κάποιου που άμεσα σχετίζονται με ε, τρομοκρατικού πυρήνε και ενδέχεται να διαπράξουν ε, τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό είναι βασικό παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα ποινικοποίηση ε, ε, μιας μη δημοφιλούς αποψη που πρέπει να διαφέρεται από την, διαφοροποιείται συγγνώμη, από την ποινικοποίηση μιας, της ίδιας της πράξης. Δηλαδή να βάλει κάποιος μια βόμβα παραδείγματος χάρη κάπου. Ε, και μπορεί να αποδειχθεί και αντιπαραγωγικό από πολιτικής άποψη. Αν πολλοί έχουν εκφράσει ριζοσπαστικές απόψεις, ε, ε, αν υποστηρίζουν δηλαδή τρομοκρατικές ενέργειε. χωρί όμως να εμπλέκονται άμεσα, μπορεί να, να γίνει πιο ριζοσπαστική λοιπόν η δράση αυτών κάποιων ομάδων και ε, ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε ε, άθελά μας ε, και διαφήμιση αυτών των ριζοσπαστικών ομάδων και δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην πρόληψη της τρομοκρατίας. Θεωρώ ότι μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγικό από πολιτικής άποψης και προβληματικό από πλευράς παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τις συμβάσει του Συμβουλίου της Ευρώπης και για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι θα υπάρξει ικανοποιητική εφαρμογή. Περνάω στα μέτρα της κοινότητα και κυρίως το θέμα της προστασίας και της διατήρησης των δεδομένων. Ε, η, νομοθεσία, η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων όπως εξάλλου ε, και η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παράνομη υποκλοπή των δεδομένων. Δεν είναι ταυτόσημα τα ζητήματα, αλλά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό επικάλυψη. Οπότε καλό θα ήταν, όπως λέω μέσα στην έκθεση, να δούμε αν η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να διευρυνθεί για την προστασία των δεδομένων, ώστε να καλύπτει και τα το ποινικό δίκαιο. Ε, δηλαδή να προβλέπεται η ε, υποχρέωση ε, να τιμωρούνται οι παραβιάσεις της, του απόρριτου χαρακτήρα των δεδομένων μέσα από το ποινικό δίκαιο όπου δει. ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό το θέμα γιατί έχουμε τη σχέση του πρώτου και του τρίτου πυλώνα συνθήκες Λισαβόνας αν επικυρωθεί θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Αν όχι, θα πρέπει παρόλα αυτά να ε, δούμε ε, πώς έχει η κατάσταση, δηλαδή να δούμε αν οι ποινικές, ε, χάρη στις ποινικές κυρώσεις θα υπάρχει ε, καλύτερη προστασία κατά της παραβίασης ε, των κανόνων, ε, κυρίως όταν μιλάμε για την παραποίηση ταυτότητας και για το phishing. Αν υπάρχουν υποχρεώσεις μέσα στο ποινικό δίκαιο, δηλαδή στο αρχικό στάδιο, όταν έγινε η υποκλοπή, όταν έγινε η παραβίαση, ίσως υπάρχει πιο αποτελεσματική προστασία. Επίσης το spam, τα ανεπιθύμητα email. Έτσι θα μπορούσαμε με πιο αποτελεσματικό να εφαρμόσουμε την νομοθεσία και συμφωνώ με τον Peter Hastings ότι υπάρχουν και δύσκολα ζητήματα ε, στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Ούτως ή άλλω η δικαιοδοσία, η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου ε, για την εφαρμογή των μέτρων ε, εντό και εκτό κυρίω Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέματα που πρέπει να μα απασχολήσουν. Το, η διατήρηση των δεδομένων, αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι σε αυτό εδώ, συμφωνώ με το σχέδιο της έκθεσης του εισηγητή ότι δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει γενικευμένη παρακολούθηση της χρήσης του ίντερνετ ε, από όλους. Απλά η οδηγία της ε, διατήρησης των δεδομένων που έχει ήδη είχε εγκριθεί προς αυτή την κατεύθυνση πάει ακριβώς και αν μας ανησυχεί ε, η πρακτική η εφαρμογή, η επίτευξη του στόχου του εισηγητή, δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι επί της αρχής ε, υπάρχει χρήση του διαδικτύου χωρίς παρακολούθηση καταρχάς, ε, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή την οδηγία διατηρήσης των δεδομένων το ταχύτερο δυνατόν, ούτως ώστε να το ρυθμίσουμε το ζήτημα και ε, συγκεκριμένα όπως ίσως γνωρίζετε, η οδηγία διατήρησης δεδομένων θα εφαρμοστεί στο διαδίκτυο σε 10 μέρες από τώρα ε, σε κράτη-μέλη που έχουν καθυστερήσει ε, με την εφαρμογή της ε, οδηγίας στο διαδίκτυο. Από 15 Μαρτίου θα αρχίσει να ισχύει. Δεν υπάρχει κανένα όριο σε σχέση με το ποιο έχει πρόσβαση σε αυτά τα διατηρηθέντα δεδομένα ε, και για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει και ανώτατη περίοδος, γιατί η σε περίοδος μπορεί να παραταθεί. Ε, και η οδηγία διατήρηση δεδομένων αφήνει ακέραιες εφεδρικές λύσεις για τα κράτη-μέλη για τη χρήση των διατηρηθέντων δεδομένων για άλλους στόχους πέρα από την δίωξη σοβαρού εγκλήματος, για πολιτικούς λόγους, για πρόληψη του εγκλήματος, ε, για δίωξη λιγότερο σοβαρών αδικημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Ποια σχέση ανάμεσα στην ε, πρόβλεψη της υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων για σκοπούς έρευνας σοβαρών εγκλημάτων ε, και των υπολείπων εναλλακτικών λύσεων. Δηλαδή, ε, μέχρι που προβλέφθηκε αυτή η δυνατότητα διατήρηση δεδομένων, κάποια κράτη-μέλη προ τα εκεί οδεύαν έτσι, σε εθνικό επίπεδο. Αλλά μέχρι που δημιουργήθηκε αυτή η υποχρέωση ε, σε κοινοτικό επίπεδο, κάποια κράτη-μέλη δεν είχαν στόχο να κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ήθελαν επίσης να επιβάλλουν το κόστος διατήρησης δεδομένων στην βιομηχανία, γιατί δεν υπήρχε κοινοτικός κανόνας ε, ε, που να εξισώνει το κόστος, δηλαδή να το κατανέμει ισότιμα ανάμεσα στο κράτος και στην εταιρεία. Τώρα όμως λήφθη η απόφαση να διατηρούνται όλα αυτά τα δεδομένα για συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων. Μα είναι κάτι υπαρκτό πλέον και το κόστος της βιομηχανίας ε, έχει επιβληθεί το κόστος ήδη στη βιομηχανία και ε, έχουμε, ε, το έχουμε κάνει αυτό το βήμα και συλλέγονται δεδομένα για το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο για τους επόπτους, ε, ε, ε, ε για σοβαρά εγκλήματα. Αυτό αποτελεί καμπή, ε, κατά τη γνώμη μου. Αλλάζει δηλαδή η ίδια η αντίληψη σε σχέση με την ιδιωτική ζωή και φυσικά είναι πολύ δελεαστικό να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα δεδομένα για άλλους στόχους, έτσι. Ε, πηγαίνετε σε ένα παιδικό πάρτι με ένα σάκο, με σακίδιο, με ε, καραμέλες και γλυκά. Και θα πείτε στα παιδιά, για κοιτάξτε τι έχω εδώ, αλλά δεν σας τα δίνω. Ε, όταν φύγετε ε, θα εξαφανιστούν, ε, ρηπεί φθαλμού, όλα, όλες καραμέλες και όλα τα γλυκά, έτσι είναι λογικό. Εάν προσπαθήσετε να τους εμποδίσετε, θα πρέπει να επιχειρηματολογείτε και να τους εμποδίζετε συνέχεια. Ε, τι εννοώ. Έχω τέσσερα μικρά παιδιά, γι' αυτό πήρα και αυτό το παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό ο παραλληλισμός για τη συλλογή των δεδομένων. Αφού υπάρχουν ναι, ε, μέσα στο σάκο τα δεδομένα, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, ε, αν ξέρουν ότι μπορούν να τα πάρουν, θα τα πάρουν. Και όσοι που ε, και θα γκρινιάζουν μέχρι να να τους δοθεί η πρόσβαση στα δεδομένα και αν φύγετε και δεν υπάρχει κλειδαριά, δεν υπάρχει δικλείδα ασφαλείας, ε, τους αφήστε μόνο στο δωμάτιο με τα δεδομένα, αν δεν χρειάζεται νομική έγκριση για την ε, χρήση αυτών των δεδομένων, ε, κάποιοι θα παρακάμψουν ε, αυτά τα, αυτούς τους κανόνες και θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Το DNA παραδείγματος χάρη των υπόπτων. Φύγανε οι καραμέλες λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν ήδη τα δεδομένα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα δεδομένα, όποιος τα θέλει θα τα πάρει, ακόμη και αν δεν υπάρχει επίσημη έγκριση. Τώρα τα κράτη συλλέγουν τα δεδομένα και βλέπετε τι γίνεται. Οι δισκογραφικές εταιρείες ε, ζητάνε να κοινοποιούνται τα δεδομένα προ τα δικαστήρια. Ε, τα κράτη-μέλη ε, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και ασκούνται σοβαρές πιέσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί κάποια κράτη-μέλη να θεωρούν ότι η βιομηχανία τους ε, η μουσική βιομηχανία δεν προστατεύεται επαρκώ, κάποια έχουν αρχίσει να ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για τη διδίωξη σοβαρών εγκλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί χρησιμοποιούνται και για άλλου ε, στόχους. Ε, για οτιδήποτε λύσει η αρμόδια αρχή να τα χρησιμοποιήσει. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή στα σοβαρά εγκλήματα επί της ουσίας και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Το 2005 δεν δεν ε, το είχαμε φανταστεί ότι θα συνέβαινε αυτό και εγώ ίδιος και άλλοι το είπανε ότι μπορεί να συμβεί αυτό τώρα, συμβαίνει ήδη. Ε, πρέπει να αναθεωρηθεί οπωσδήποτε η οδηγία διατήρησης ε, των δεδομένων και να ενισχύσουμε τους στόχους του σχεδίου συστάσεων γιατί υπάρχει μαζική παρακολούθηση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Αυτά και με χαρά να απαντήσω και σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε, αυτές είναι βασικές ανησυχίες ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως προς την ανάγκη να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν υψηλότερα πρότυπα για το κυβερνό έγκλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. For, ε, for a couple of minutes... Σας ευχαριστώ πράγματι. Συζητούσαμε τη γραμματεία και σχολιάζαμε το πόσο συναρπαστική είναι αυτή η ακρόαση και πόσο πολύτιμη είναι κάθε παρέμβαση και συζητούσαμε αν είναι δυνατόν να έχουμε τα πρακτικά και να τα μοιράσουμε στους βουλευτές και σε οποιονδήποτε άλλον θέλει. Πριν περάσουμε στην φάση των τελευταίων παρατηρήσεων. όποιο θέλει να κάνει κάποιε ερωτήσει να συζητήσουμε κάτι, αν έχετε κάτι να πείτε, ε, τώρα είναι η στιγμή να λάβετε τον λόγο. Και εκτός βεβαίως αν έχετε μείνει άναυδοι από την ποιότητα των παρουσιάσεων και δεν τολμάτε να κάνετε καμία ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σκεφτείτε κάποια ερώτηση, να απαντήσω εγώ σε μια ερώτηση του Γκράσα για το παράγραφο στην ερώτησή μου για διατήρηση δεδομένων. Οπωσδήποτε κάτι αναφέρεται, αλλά δεν, δεν το λέμε ανοιχτά. Εγώ προσωπικά είμαι, ήμουν κατά αυτής της οδηγίας και ήμουν ε, μειονότητα τότε βεβαίως, αλλά να είμαστε και δίκαιοι με το Κοινοβούλιο για την διατήρηση των δεδομένων. Ήταν ε, περίεργες εποχές. Ε, η Βρετανική Προεδρία ήρθε και είπε στο Κοινοβούλιο πως παρά το ότι εγώ πιστεύω ότι δεν έχετε απόφαση και παρά το ότι και πολλοί άλλοι πρωθυπουργοί πιστεύουν ότι δεν έχετε θα σας κάνω τη χάρη να δούμε αυτό το ζήτημα σαν να είχαμε στην απόφαση. Οπότε πολλοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι αυτό ήταν το άνοιγμα της πόρτας για την απόφαση στον τρίτο πυλώνα μέσω της ε, λεγόμενης αυτής ρήτρας πασαρέλας. Μπορεί να μην σα λέει τίποτα αυτή η συζήτηση, αλλά διαδικαστικά είναι πάρα πολύ σημαντική μέχρι να έρθει η συνθήκη τη λισαβόνα ενισχύει. Δεν έχει συναπόφαση, δικαίωμα τη συναπόφασης το Κοινοβούλιο για ζητήματα τρίτου πυλώνα, δηλαδή αστυνομική συνεργασία κτλ. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή τη οδηγία ήταν πώς υπάρχει η χρειά που έδωσαν πολλές κυβερνήσεις, αστυνομική τα λοιπά. Γιατί το αναφέρω αυτό. Μιλάμε για δεδομένα ιδιωτών που συλλέγουν ιδιωτικές εταιρείες για τους ιδιωτικούς τους σκοπούς. Π.χ. εταιρείες τηλεφωνικές ε, για να στέλνουν σωστά τους λογαριασμούς και διατηρούνται αυτά για όσο καιρό θεωρούν σωστό οι εταιρείε αυτές. Οπότε η όλη διαδικασία της διατήρησης δεδομένων όπως ξεκίνησε και συνέβη με τις εταιρείε, γιατί έγινε αυτό, ήταν ξεκάθαρα ιδιωτική. Δηλαδή 95-46 πρώτος πυλώνας αυστηρά. Και ξαφνικά οι κυβερνήσεις λένε «Α, θέμε κι εμείς» για τους δικούς μας σκοπούς και έτεθη μετά ένα πολύ ενδιαφέρον νομικό ζήτημα. Δηλαδή, λέγοντας μόνο ότι ο σκοπό μα είναι τρομοκρατία, κάτι τελείως ιδιωτικό, το αντιμετωπίζουμε μέσω ενός τελείω διαφορετικού νομικού συστήματος τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Το ΔΕΚ στην ε, διαβόητη υπόθεση PNR ψυχείων ε, αεροπορικών επιβατών εξέδωσε μια γνωμοδότηση πολύ ανησυχητική κατά την άποψή μου. Κατ' ουσίαν είπε πως όταν οι αεροπορικές εταιρείες συλλέγουν δεδομένα ε, προσωπικά δεδομένα επιβατών για τους σκοπούς τους, δηλαδή για να σου την κράτηση, ξέρω εγώ. Εφή στιγμή που ένα κράτος δηλώνει, ούτε καν ευρωπαϊκό, τρίτο κράτος ζητάει αυτά τα δεδομένα για λόγους ασφαλείας, γίνεται αυτό τρίτος πυλώνας. Δηλαδή έδωσε το δικαστήριο σε μη κράτος μέλος να ορίσει τι θα γίνουν τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας τρίτη χώρα έτσι ότι τα θέλει για τον χύψη σκοπό. Πολύ περίεργη απόφαση. Αλλά αυτή ήταν. Λοιπόν, προσπάθησα να τραβήξω όσο μπορούσα ε, για να σκεφτείτε κάποια ερώτηση. Αλλά πέραν όχι, θα περάσουμε φαντάζομαι στα συμπεράσματα. Λίγο νωρίτερα μάλιστα από ό,τι περιμέναμε. Ο κύριος Πελτομάκη είναι εδώ. Ωραιότατα. Και ο κύριος Βαζέλσκι είναι απ' έξω, μάλιστα. Νομίζω πως θα ευχαριστήσω εδώ τους ομιλητές μας ε, για την παρέμβαση αυτή. Οπωσδήποτε θα συγκεντρώσουμε τα πρακτικά